εβδομάδα εστιάζω την προσοχή μου στα θέματα που αφαιρούν άμεσα τη δική μας Επιτροπή. Λοιπόν, θα αρχίσω χαιρετίζοντας ε, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, διότι πρόκειται για την σφαιρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μεταναστευτικά ζητήματα. Ε, υπάρχουν τα απαιτούμενα ε, μέσα ως προς το προσωπικό και τα οικονομικά μέσα για να ε, ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτού του ζητήματος. Ολιστική λέγεται η προσέγγιση, κύριε Ντεπρέ. Έτσι τη λένε, τι να κάνουμε. Είπε, είπα ότι χαιρετίζω την, το σχέδιο διότι ε, υπάρχουν τα πετούμενα μέσα για την υλοποίηση του σχεδίου. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, αμφιβολίες ή ε, είναι και εχθρικά σε σχέση με δύο δράσεις ε, για την μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων για ένα συνολικό ποσό 240 εκατομμυρίων και στη συνέχεια την επανεγκατάσταση 20.000 ατόμων για ένα ποσό 120 εκατομμυρίων από το Ιράκ. Δεύτερον, προτείνεται αύξηση για το 2016 για το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρόκειται για μια αύξηση 202 περίπου εκατομμυρίων και ο συνολικός προϋπολογισμός 200.000. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μία αξιολόγηση των αναγκών για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, ε, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε ταχύτατα ε, στις ενδεχόμενες προτάσεις για αύξηση των κονδυλίων στα πλαίσια της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών. Είμαι πεπισμένος ε, ότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε σε αυτά τα προβλήματα που μας εξέδεσε ο κ. Λιτζέρη για, τα, για τις μεταναστευτικές επιέσεις, τα προσεχή έχει έτη τουλάχιστον μέχρι το πέρασε του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου αν δεν υπάρξουν οι αυξήσεις λάμβανω γνώση επίσης των αυξημένων κονδυλίων για τον Frontex και ζητώ δύο πράγματα. Ε, να έχουμε επιπρόσθετο προσωπικό, τόσο ώστε να υλοποιούνται αυτές οι επιχειρηματικές δράσεις του Frontex και ζητάμε περισσότερες πληροφορίες από πλευρές Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την τροποποιημένη εντολή του Frontex για τις επιστροφές. Θα ήθελα να ε, ενημερώσω τους συναδέλφους ότι στα πλαίσια του προϋπολογισμού που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γραμμή ε, που σχετίζεται με την νόμιμη μετανάστευση και την ενσωμάτωση των επικών τρίτων χωρών ε, αλλά και σε σχέση με την ε, πολιτική επιστροφή μειώνεται σε σχέση με το 2015. Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αν είναι συνεχτική η πολιτική της. Επίσης ενισχυμένος ρόλος του ΕΑΖΟ μας τα είπε ο κ. Λιτζέρη Χρειάζεται εναρμόνιση και νομολογία κυρίως για την ταυτοποίηση των ετούντων άσυλο ως προς όλες τις διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν αλλά ταυτόχρονα και ως προς τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να χορηγηθεί ή όχι ε, το άσυλο. Υπάρχουν ε, απαράδεκτες διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, διότι ε, υπάρχουν άνθρωποι που σε ένα κάτω μέλος δεν έχουν ούτε μία στις δέκα δυνατότητα να αποκτήσουν το άσυλο, ενώ σε άλλες έχουν κάθε πιθανότητα. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι, κύριε Ντύπρε. Ε, γίνεται να περάσουν σε ένα άλλο κράτο μέρο λοιπόν και να ζητήσουν το άσυλο. Μα όχι, αυτό, περί αυτού πρόκειται στο Δουβλίνο 3. Τι γίνεται, συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πρώτο κράτο μέρο, τα είπατε και με τον κύριο Λιζέρη, υπάρχει απόπειρα ταυτοποίηση ε, του μετανάστη, ούτω ώστε να συγκροτηθεί και η βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων, Eurodac. Όταν λοιπόν ζητείτε Mm. το άσυλο σε κάποιο κράτος μέλος γίνεται έρευνα στην βάση Eurodac για να δούμε ε, αν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα και άρα αν έχει μπει ήδη και έχει προσπαθήσει να αποκτήσει άσυλο σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Αν διαπιστωθεί ότι αυτό έχει συμβεί πρέπει να επιστραφεί ε, ο άνθρωπος αυτός στο κράτος μέλος όπου έχει κατατεθεί η πρώτη αίτηση ασύλου. Επίση, δεν πρέπει να έχουμε αυτόματες και γραμμικές μειώσεις, ε, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τις επιχειρηματικέ ανάγκες ε, των υπηρεσιών που συνεργάζονται στα πλαίσια των hotspots ε, για τις μακροπρόθεσμες πολιτικές, ε, διότι ο κύριος Λιτζέρη μας μίλησε για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για όλες τις επιχειρηματικές δράσεις ε, από πλευράς δημοσιονομικής αλλά και από πλευράς ε, προσωπικού. Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω στους συναδέλφους μου για τα στοιχεία που θα συμπεριλάβω στην έκθεση προς νομοδότηση που θα καταθέσω την επόμενη εβδομάδα και περιμένω τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ντιπρέ ε, ήσασταν ε, συνοπτικός αλλά και διαφωτιστικός. Έτσι, ε, ε, συνεχίζουμε ουσιαστικά τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Λιζέρη. Σα ευχαριστούμε για τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την Επιτροπή Προπολογισμού. Ορισμένε φορέ ε, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ο κύριος Λαβία τώρα θα πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Il tema della situazione del Mediterraneo è un tema oggi estremamente το πρόβλημα αυτό των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο είναι πάρα πολύ καυτό σήμερα και πάρα πολύ ε, σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το ζούνε, το ζούνε με, με, όλη την αγωνία που αρμόζει όλες οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Εγώ βρέχομαι από την ε, Σικελία και η Σικελία είναι το πρώτο λιμάνι στόχος, προορισμός τέλο πάντων σε αυτή τη φάση της μετανάστευσης και η κατάσταση τη, μία μέρα μετά την άλλη γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη και όλο ένα και περισσότερο ε, ε γίνεται πήγον το να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν επομένω ε, το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί μόνο από τι χώρε που βρίσκονται στα σύνορα τη κοινότητα. Βέβαια, τώρα μιλούμε για τον προπολογισμό και σα παραπέμπω σε αυτά τα οποία ε, αναφέρθηκαν προηγουμένω. Γιατί δεν μιλούμε τώρα για κάτι το ευκαιριακό, κάτι το σημειακό. Μιλάμε για μια ολόκληρη διαδικασία, μια ολόκληρη πορεία που έχει κρατήσει κάποια χρόνια και θα κρατήσει και άλλα. Οπότε και αυτό με, με να σας πω ότι από πλευράς δημοσιονομικής, πλευράς προϋπολογισμού δεν είναι εύκολο έτσι να λυθεί το πρόβλημα γιατί δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας των χώρων αλλά κυρίως διότι τώρα μιλούμε για μια καινούρια ανάπτυξη, για μια επαναχρησιμοποίηση των κονδυλίων του προπολογισμού. Μιλάμε τώρα για μια τέτοια πορεία μετανάστευση, ε, μια εξέλιξη στη μετανάστευση που κρατάει τόσα χρόνια και πρέπει από εκείνο να αντιμετωπίσουμε γιατί ακόμα και για τη χρήση του 2017 θα πρέπει να δούμε αν υπαρκούν τα κονδύλια και άρα αυτό να κάτσουμε να σκεφτούμε γιατί ήδη το Συμβούλιο ε, είπε και έκρινε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα θεματολόγιο και να έχουμε κάπου καταγεγραμμένα τα σημεία εσόδου, τα hot spots. Μια που ξαναμιλούμε για αυτήν την ε, ε, κατανομή αυτών των 40.000 ε, μεταναστών που φτάνουν πέρα από το Κύρκο, μόνο 5.000 έρχονται στην ε, Σεκελία, ξέρετε. Άρα το θέμα που τώρα πια άλλες διαστάσεις. Άρα θα πρέπει και συνδυασμό με την Επιτροπή Λίμπε να δούμε τι θα κάνουμε. Είτε απίστευτες οι διαστάσεις του θέματος και γι' αυτό σας λέω ότι και από πλασδί μισονομικής θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή πορείας και θα πρέπει να ληφθούν κάποια επιπρόσθετα μέτρα και ακριβώς να δούμε τι γίνεται με τα hot spot, να δούμε πώς θα έχουμε ε, κάποιο είδους ειδικέ δομές για την ε, πρώτη υποδοχή των ανθρώπων αυτών. Άρα και δημεσονικά να κάνουμε μια στροφή και να έχουμε κάποια ειδικά κονδύλια. Και ακριβώς να υπάρχουν τα χρήματα που χρειάζονται και να μην γίνεται επιστροφή, ανάκτησή τους. Κάτι άλλο τώρα. Έχουμε τώρα μπροστά μας ε, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αυξάνονται οι ροές μεταναστευτικέ. μεταναστευτικές. Επομένως ακόμη περισσότερο χρειάζεται να ενεργήσει, να κάνει κάτι η Ευρώπη στα σύνορα. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Τα λέμε στην Κατάνια. Επειδή έχει περάσει η ώρα, ε, καλύτερα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν πάντοτε ζητήματα. αλλά ούτως ή άλλως είναι ένα από τα ζητήματα που θα πας αποσχολήσουν ε, στο μέλλον. Ε, υπάρχει έκρηξη στη μεταστευτική πίεση όπως είδαμε και από τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία μας έδωσε ο κύριος Λιτζέρη. Λοιπόν, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θα ήθελα να σας κοινοποιήσω τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές ε, στις 8 Ιουνίου ε, αποφάσισαν να καταθέσουν γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση 2014 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η ε, κυρία Γωνία Ζαμπάλ θα υποβάλει την αναφορά. Στη συνέχεια θα ε, καταθέσουμε γνωμοδότηση για την, το θέμα της διεθνούς προστασίας ε, ως ως την Ιταλία και τη Γαλλία. Πάλι βλέπετε τα προβλήματα της μεταναστευτικής πίεσης. Ε, το ΕΛΚΑ είχε αναλάβει αυτή τη γνωμοδότηση και τελικά... Λαμβάνοντα υπόψη το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα εργασία, σήμερα το πρωί συμφωνήσαμε ο υποφαινόμενο να ε, στείλει μία επιστολή στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για αυτό το θέμα προβλέπεται να συντάξουμε έκθεση για την κινητοποίηση των ε, μέσων ευελιξίας για τη διεθνή προστασία πάλι ε, προς όφελος της Ιταλίας ε, και της Ελλάδας. Ο Χουσέ Μανουέλ Φερνάντες είναι ο εισηγητής. Επίσης θα συνταχθεί έκθεση για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης για την καταβολή προκαταβολών ναι, για την προϋπολογισμό του 2016. Ο κ. Χριστοφόρου είναι ο εισηγητής ε, εξ του ΕΛΚ. 16 Ιουνίου οι συντονιστές ε, σε μια έκτακτη σύσκεψή τους ε, αποφάσισαν την δίκαιη κατανομή των μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Επιτροπής Προϋπολογισμών στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στη Σικελία τον Ιούνιο και αποφάσισαν 8 μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών και 4 μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να ε, συμμετάσχουν στην αποστολή αυτή. Και επειδή υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για αυτή την αντιπροσωπεία, ε, ε, είναι δυνατόν να, υπάρξουν, ε, ε, να υπάρξει ένας διπλάσιος αριθμός μελών, 12 μόνιμα μέλη και 12 συνοδευτικά. Ελπίζουμε ε, να συμφωνήσουν τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του διαρθρωμένου, ετησίου διαρθρωμένου διαλόγου, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της όλου ιδιαίτερως στην αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγράψει αυτό το στόχο της αναθεώρησης στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016. Εκφράσαμε επίσης την επιθυμία μας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας διαφωτίσει ως προς τις ικανότητες απορρόφησης και χρήσης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς των κρατών μελών, μιλώντας κυρίως για τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Επίσης, μία ειδική αποστολή για τις προοπτικές των πληρωμών και των ανεξόφλητων λογαριασμών μέχρι το πέρασε του δημοσιονομικού πλαισίου ε, μας έκανε μία αναισθητική ένεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι μας, είπε, μας μίλησε για τα 2 δις το 2016 όμως μην ξεχνάμε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο πάει μέχρι το 2013 και ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να συσσωρευτούν και πάλι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ε, ε, στο πέρας του τρέχοντος ε, δημοσιονομικού πλαισίου κατόπιν για τα ειδικά ταμεία και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εξακριβώσουμε ότι για τους ειδικού οργανισμούς δεν ε, υπάρχει πλήρη σεβασμός των πρωταρχικών στόχων των οργανισμών. Οι συντονιστές επίσης ενέκριναν δύο σχέδια επιστολών ε, που συνέταξα. Ε, ε, μία επιστολή προς τον Αντώνιο Παντσέρη, τον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων των αντιπροσωπιών, το είπα, το κατάφερα. το αντικείμενο είναι να βελτιώσουμε το συντονισμό των συναρμοδίων επιτροπών και των αντιπροσωπιών. Και επίσης ε, μία επιστολή του συναδέλφου Πατριτσέλο που ζήτησε ένα ειδικό ταμείο για να καλυφθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί διάφορα κράτη-μέλη από το εμπάρκο ε, που έχει επιβληθεί κατά της Ρωσίας. Ιδού, σας ενημέρωσα για όλα τα ζητήματα και θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να βάλετε την ε, κάρτα ψηφοφορίας ε, στα ειδικά μηχανήματα για να κάνουμε μια δοκιμή. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34 προς 36 ε, δεν έχουν ψηφίσει δύο ενώ είχαμε τις κάρτες 35 άλλη μία ψήφος μας λείπει ελέγξτε παρακαλώ μήπως υπάρχει ένα μηχάνημα που ε, δεν ε, χρησιμοποιείται όχι Έχουν λάβει όλα τα μέτρα τους, τι να πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έκθεση του Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες για την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Κύριε Μπέγκε. Συντομότατα, <clears throat> η κυρία Χολμάερ και εγώ έχουμε καταθέσει τροπολογίες 41 και 42 για το ΙΤΕΡ και για το εξωτερικό εργαλείο χρηματοδότησης. Θέλουμε να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε προβλήματα. Για αυτές τις τρεις τροπολογίες τις αποσύρουμε, αλλά για το ίτερ θέλω να τονίσω ότι το θέμα της έγκαιρης παράδοσης αναφορών για το ίτερ παραμένει ένα σημαντικό θέμα και εμείς πιστεύουμε πρέπει να σκεφτούμε για ένα αποθεματικό για να δείξουμε τις επιφυλάξεις μας και επίσης και για το εξωτερικό εργαλείο χρηματοδότηση υπήρξαν κάποιες εντάσεις. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό πάλι με ένα αποθεματικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξει αυτό το εργαλείο, να αντιμετωπιστεί πιο προσεκτικά και να σκεφτούμε καλύτερα για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να πάρει αυτό το εργαλείο και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας φύγει, να μας ξεφύγει αυτή η ευκαιρία για μια πιο μεγαλύτερη σαφήνεια για αυτό το εργαλείο στη διαδικασία του προπολογισμού. Αποσύρουμε πάντως τις τροπολογίες μας για να μην επιβαλύνουμε τη διαδικασία. Η κυρία Χολμάια. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο ε, Μπέγκε για το ΙΤΕΡ. Θα έρθει η έκθεση αυτή τον Ιούνιο και τώρα δεν ξέρω πού θα θέλουμε να έχουμε τις πληροφορίες για τις εκθέσεις αυτές αλλά νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει ήδη ότι δεν θέλουμε να επαναφέρουμε ε, τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν του Σεπτέμβριο γι' αυτό είναι απαραίτητο η έκθεση αυτή να είναι οπωσδήποτε διαθέσιμη το Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες στον προπολογισμό μα, γιατί αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αποδεκτά. Το σημειώνουμε. Λοιπόν, αποσύρεται τι 40, 41, 42, 43 τροπολογίες. Σωστά. 41, 42, 43. Δεν είναι μέσα μια συμβαστική αυτές. 41, 42 δεν καλύπτονται από τη συμβαστική ε. 47, 73, 73 λέτε. Και λοιπόν ποια είναι η τύχη τώρα πλέον του... τη συμβαστική ε. Α, όχι, κατέπιπταν. Ακριβώ επειδή υπήρχε η συμβαστική. Οκ. Λοιπόν, παράγραφος 1, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 για την παράγραφο 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Είναι με προφορική τροπολογία. Πιστεύει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα ώστε να βοηθήσουν τα κρατη μελέτη να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως με απώλεια ανταγωνισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 με προφορική τροπολογία λόγω της αυξανόμενης πίεσης των μεταναστευτικών ρόλων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 με προφορική τροπολογία θα ε, δώσει ιδιαίτερη σημασία στην κινητικότητα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταπευθούν οι 12, 13 και 14. Η συμβαστική β. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται παράγραφος 6 τροπολογία 18 υπέρ αν έχει προφορική τροπολογία Regrets of criticism υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Mm. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα με προφορική τροπολογία and accounting for inflation μέχρι το real terms. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα με μια προφορική τροπολογία που αποδίδει έμφαση στην σημασία της αποτελεσματικότητας ε, της, ε, των δαπανών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολο... Ε, παράγραφος 10α, ναι, τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταπίπτουν 20, 27, 30 και 34. 12 ε, ε, η τροπολογία 31 με προφορική τροπολογία δυνάμει του άρθρου 310 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δαπάνες και τα εισοδήματα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ισορροπημένα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Προφορική τροπολογία. Μέχρι τα προγράμματα συνοχής. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 33. Υπέρ. Κατά. Έχουμε και προφορική τροπολογία πρέπει να πάει στην παράγραφο 41 κτλ. κτλ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική δέλτα για την παράγραφο 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και καταπίπτουν οι 28, 35 και 36 που καλύπτονται από αυτήν. Παράγραφος 16 έχει αποσυρθεί η τροπολογία. Για τη 16α έχουμε τροπολογία 38. Προφορική τροπολογία εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αντικτύπων ως προς τη χρηματοδότηση έρευνας για το κλίμα, τις κλιματικές αλλαγές, για την επιστήμη στην κοινωνία κτλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σημαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 44 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική F παράγραφος 21 τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 21, τροπολογία 50, υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 49 λέει ο πρόεδρος και τώρα θα διορθώσουμε μάλλον. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος 50 ε, για την παράγραφο 21α, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, η τροπολογία 51 για την παράγραφο 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, 22 συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 22α, τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23 υπέρ. τροπολογία 56 υπέρ. Ναι. εκτός παιδίου και μη παραδεκτή τροπολογία 26α, τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Έχουμε και προφορική τροπολογία για, που λέει την προσθήκη της πρότασης παράγραφο 26. Ποιος είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας 57, της τροπολογίας 57 με την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Για πάμε τώρα στην παράγραφο 28. H. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 29 ή 66 είπε. Κατά. Θα κάνουμε μια επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 31 ή 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 68 με μια προφορική τροπολογία πιστεύει ότι περαιτέρω ενίσχυση κάποιων ζωνών προτεραιότητες όπως η Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και η αρρωγή προς την ειρευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής για την Παλαιστίνη και για την αποστολή του ΟΗΕ θα χρειαστεί λόγω της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Ε, ε, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. Παράγωση 32, τροπολογία 69, υπέρ. Κατά. Απόχες. Απολύτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 έχει αποσυρθεί 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 με προφορική τροποποίηση including initiatives aimed at reflecting and accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική εν ή υπέρ κατά αποχές γίνεται δεκτή συμβαστική αι αιτιολογικές αναφορές Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γνωμοδοτήσεις τώρα των επιμέρους επιτροπών. οι περισσότερες τροπολογίες καλύπτονται ή είναι εκτός πεδίου τροποποίησης. Η πρώτη τροπολογία πρέπει που να αντιμετωπίσουμε είναι η EMPL 3, τροπολογία 3 της Επιτροπής Απασχόλησης, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. EMPL 6, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 9 ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία της Επιτροπής ε, Άγκρη. Άγκρη 19. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλία ΠΕΣ 6 με προφορική τροποποίηση including the, through the collection of data υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην Επιτροπή Προ... Πολιτισμού Κουλτ 1 με προφορική τροποποίηση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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών ΦΕΜ 2 Τροπολογία 2 Προφορική Τροποποίηση Recalls that the issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση όπως έχει τρομοποιηθεί. άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική κλίση ψηφίσατε όλοι λείπουνε δύο εντάξει πέρας εγκρίθηκε η εντολή του κυρίου Φερνάντες 29 υπέρ, 4 ψήφι κατά, 4 αποχέ. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 1 που παρουσιάζεται από την κυρία Γουάρδια Σαάλ. Έχετε εδώ μία σειρά από τροπολογίες. Υπαριθμόν 1 πρώτα. Εντάξει κυρία Σιγητρία. Διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 1. Έχετε λοιπόν μία σειρά τροπολογιών που θα ψηφιστούν σε μπλοκ. Η εισηγήτρια έχει αρνητική άποψη. Συμφωνείτε για να έχετε μία ομαδική ψηφοφορία. Ναι. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται αυτές τις τροπολογίες. Και τώρα ψηφίσουμε την έκθεση για το διορθωτικό προϋπολογισμό, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Είναι συμβατή με την 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση στην 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται στο τσακ. 17-18. Τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη σε. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι γνωμοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών καλύπτονται όλες για την Ήτρε, για την Τραν, παράγραφος 2. Μια προφορική τροποποίηση επενδύσει στην έρευνα και τη μεταφορά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτσι, στην παράγραφο 2. για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού συνεργειών μεταξύ του ΕΣΥΦ και του ΕΦΣΥ ενώ ενισχύει και πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται με 27 υπέρ εναντίον 5 και με 5 αποχές. Υπαριθμόν 3. Διορθωτικός προϋπολογισμός. που αφορά το πλεόνασμα του έτους 2014. Έκθεση της κυρίας Γουαρδιά Σαβάλ. Η 1 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 2 της υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι τροπολογίε 3 και 4 έχουν αποσυρθεί. Το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 1 αποχή. διορθωτικός προϋπολογισμός 4 για το 2015 για την κινητοποίηση, την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία. Έχει αποστεί το, η τροπολογία 2, το, η 3, ε, με την προφορική τροπολογία. Λέμε το, λαμβάνει υπόψη ότι το Ταμείο για την Ελληνική θα πρέπει να δείξει ελληνική με τον κόσμο ή στην περιοχή που επλήγει από τις θεομηνίες. Υπέρ, κατά. Αποχές. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Considérant 1, amendement numéro. Ε, παράγραφος Α. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα για το, για το σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Manque deux votants. Άλλοι δύο, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους, ε, μία ψήφος κατά και πέντε αποχές. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία για την έκθεση κ. Μιρέσαν Τροπολογία 3 για την παραγραφό 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 προς 15 και μία αποχή. Η παράγραφος 1α, τροπολογία 4, είπε. κατα Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1α, τροπολογία, φοροφορική τροπολογία. Involving by examining, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Καταπίπτει, λέει εδώ, να εγκρίνεται, αν είχε εγκριθεί η πρώτη τροπολογία, είχε απορριφθεί όμως, οπότε ψηφίζουμε για αυτήν υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Technical change λέει εδώ. Ε, για την αιτιολογική σκέψη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 2, τεχνική αλλαγή επίσης υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται και το, το τροποποιηθέν κείμενο θα το ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. 35 ψήφοι υπέρ. Καμία κατά, δύο εποχές. Τώρα, ε, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 5 για το 2015 για να ανταποκριθούμε στις μεταναστευτικές πιέσεις. Πρόκειται για τη συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε αρχίζοντας την απογευματή μας συνεδρίαση. Γκαρδία Ζαμπάλ Ρουμπιάλ. Λοιπόν, τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγουσα 3, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 για την παραγράφο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 παράγραφος 4 με χωριστή τροπολογία, ε, με ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα τονίζει μέχρι τη διαφάνεια. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Το υπόλοιπο. Υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε μία επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4α με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 14 και 15 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 5 καλύπτεται. Η 6 με μια προφορική τροπολογία whereas if migration flows are not managed in an effective and timely manner they may lead to considerable costs. Είναι πολύ serious. Υπέρ. Κάτα. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα. Οι τροπολογίες που αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Πρώτη παράγραφος. Καλύπτεται. Δεύτερη παράγραφος. Ποιοι είναι υπέρ. Α, θα πρέπει να ψηφιστούν όλες μαζί. Ωραία, το σύνολο λεγόμενων τροπολογιών της ε, ΛΥΜΠΕ. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. Για το σύνολο του, του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32, 3 και 2 αποχές. Κινητοποίηση του Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Φιλανδία. Τρία. Παρα... Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγραφός 4. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά να κάνουμε επαλήθευση. Είναι η τροπολογία 5. Σκοτάει Είναι approuvé. Ah Εγκρίνεται. Α, 18-18 ισοψηφία. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει απόρριψη, μάλιστα. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Qui s'abstient, il est Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για την τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ε, 16-20, άρα απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας και εγκρίνεται 31-5. Και τώρα. Ε, ταμείο και ταμείο επενδύσεων και χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Πρόκειται για την έκθεση Λεβαντόφσκη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία υπαριθμών 2 καταπίπτει διότι υπαριθμόν 1 εγκρίθηκε. Αλλά δεν εγκρίθηκε. Άρα, λέει ο πρόεδρος, επομένως πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά. Μάλλον ε, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμόν 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγράφος 3. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Κάνουμε επαλήθευση του αποτελέσματος ψηφοφορίας για το 8. Πέρας. Και απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 αποσύρεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 παράγραφος, τροπολογία 17, υπέρ κατά. Α, αποχές. Α, απορρίπτεται. Όχι, καταπίπτει. λέει ο πρόεδρος, συμπαθάτε με. Τροπολογία 18. Επίσης ε, καταπίπτει, όπως επίσης και η 19. Συμβαστική υπερθμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εδώ έχουμε τη συμβαστική υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 3. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 22. Α, καταπίπτει, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε της 18, 7, 12 αποχές και εγκρίνεται. Και τώρα... Α, έχω ακόμα ένα κείμενο. Α, ah oui. moi Το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Γουινέα Μπισάου. Θέλει κάποιος το λόγο. Όχι. Τότε, τροπολογία είναι υπέρ. Κάτα. Όχι, ούτε αποχές. Και... Για την έγκριση αυτού του πρωτοκόλλου ε, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Α, να ψηφίσουμε το σύνολο με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρας. 31 ψήφοι προς 2 και 4 αποχές εγκρίνεται. Για πάμε τώρα. Ε, στη μεταφορά προτείνει η κυρία Γκόρτια Ζαμπάλ. 15, 18 και 19 unblock να ψηφίσουμε. Ναι, ψηφίζουμε όμω. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για τις τρεις. Μαζί. Όλους μαζί. Αυτό είναι άμεση απόρρια της προηγούμενης ψηφοφορίας. Τρεις ε, έχουμε που δεν ψήφισαν. Δεν θέλουν ίσως. Πέρασε. 30 προς 2 και 2 εποχές εγκρίνεται. Η κυρία Σε ό,τι αφορά το DPS, είχαμε δυσκολία με τη φυσιολογική διαδικασία προκήρυξης ε, διαγωνισμού, γιατί δεν έχουν οι υποψήφοι τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνες Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μια μεταφορά πιστώσεων 10.000 ευρώ για να μπορέσουμε να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό με τη διαδικασία των contract staff, δηλαδή με άτομα επί συμβολέου. Ωραία, τότε πρέπει να ψηφίσουμε με, ονομαστική ψηφοφορία. Είναι υπέρ η κυρία Χολμάια. Παρακαλώ. Normalement, deux personnes n'ont pas encore voté. Δεν έχουν ψηφίσει δύο. Définitivement renoncé à voter. Donc... Αυτοί έχουν σταματήσει αυτοί οι δύο να ψηφίζουν εδώ και ώρα. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται 28 ψήφοι προς 3, 4 ε, αποχές. Ε, η PCA 2015, 2015, τι, αναβάλλεται αυτό, ωραία. Ε, και για Το SP Building ε, για το κτίριο είπαμε, βάλετε Για το κτίριο Άσπερ. Λοιπόν, ωραία. Ε, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Και για να ανταμυφθούμε θα ακούσουμε την πρόεδρο Γκρέσλι Για το σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού κατέληξε ο τρίλογος. Η συγγήτριά μας, η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι που μαζί με τη Λεπτονική Προεδρία, η οποία διαπραγματεύτηκε πολύ καλά και μαζί με την Κομισιόν, μπορέσαμε να κλείσουμε τον ε, τριγωνικό διάλογο. Η κατάσταση είναι ότι δεν έχουν εκφράσει άποψη στα κράτη-μέλη το σύνολο των κατών θέση για τις τροπολογίες μας. Έχουμε αναβάλει τον επόμενο τριγωνικό διάλογο, αλλά έχουμε επεξεργαστεί το κείμενο και έχουμε καταφέρει το 75% των προτάσεών μας να τις ε, περάσουμε. Και μπορώ να σας διαβάσω τώρα τι έχουμε. Έχουμε μια εξομοίωση των μη κυβερνητικών οργανισμών με τους κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτό είναι μια συμβιβαστική λύση. Εμείς θέλαμε να διαγραφεί το σημείο αυτό, αλλά η Κομισιόν θέλει να διατηρήσει αυτή την ευκαιρία της εξομοίωσης. Και έχουμε ζητήσει επίσης να υπάρξει μια εξομοίωση με σε κυβερνητικούς οργανισμούς και επίσης έχουμε εγκρίνει την άποψη για τις ε, αποκεντρωμένους φορείς. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να περάσουμε αυτές τις συμφωνίες. Έχουμε επίσης στις αιτήσει εκθέσει των Γενικών Διευθυντών μια ενισχυμένη παροχή αναφορών σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και μια μεγαλύτερη έμφαση στην προσθέμενη αξία και επίσης αυτό είναι κάτι το οποίο έχει, έχει τονιστεί από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό θεωρήθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό από το ε, Συμβούλιο, αλλά τελικά μπόρεσε να περάσει δική μας θέση. Και επίσης στις διαδικασίες προκηρύξεων διαγωνισμών να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Να μπορούν πια και οι οδηγίε μα να εφαρμόζονται και στις Βρυξέλλες και όχι μόνο στα κρατη δηλαδή. Και έχουμε τονίσει να υπάρχουν ε, καλύτερες διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις να, σε περιπτώσεις αποκλεισμού από διαγωνισμούς και επίσης ε, ζητήσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με την αναλογικότητα και την περίπτωση να υπάρξει αποκλεισμός κάποιων εταιριών και φυσικά να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου που να προσπίσει και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο σαφείς πια οι κανόνες σε σχέση με τις εξαιρέσεις και τις κυρώσεις και προτάσεις του Συμβουλίου οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την τελική απόφαση για τις ε, κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται. Υπάρχει ένα πάνελ το οποίο θα πρέπει να γίνει ακουστό σε τέτοια θέματα και μόνο σε περιπτώσεις αιτιολογημένες μπορεί να αποκλίνει ο αρμόδιος φορέας από τις αποφάσεις του πάνελ. Το πάνελ θα πρέπει να συγκαλείται όταν υπάρχει, όταν επίκειται μια σημαντική απόφαση σε διοικητικό επίπεδο. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται και να ξέρουμε αν υπάρχει μια καλή λύση. Επίσης υπάρχει το θέμα της δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Βρέθηκε μια ισορροπία η οποία για μένα εξασφαλίζει και την προστασία των δεδομένων και τη διαφάνεια. Τα νομικά πρόσωπα λοιπόν ε, καλύπτονται και οι προσωπικές εταιρείες. Εξασφαλίζουμε λοιπόν και την συνέχεια και την ε, ανεξαρτησία του πάνελ με ένα επικεφαλής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου και υψηλού επίπεδου και ανεξάρτητος και με μια γραμματεία υψηλού επίπεδου. Αυτό ήταν αίτηση του Κοινοβουλίου. Έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων όπως έχει ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε εξασφαλίσει ότι για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αντίθετα με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, να οδηγεί η μη καταβολή κοινωνικών εισφορών σε αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς. Επίσης, έχουμε κάνει μια συμβαστική λύση επί τη βάση της ειδική έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου έχουμε μειώσει το χρόνο για την καταντιμολία διαδικασία έξι εβδομάδες και τρεις ε, μήνες για το ελεκτικό συνέδριο και έχουμε προχωρήσει λοιπόν για να έχουμε μια πιο ταχεία παράδοση εκδέσεων γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάσει και μέχρι τους 20 μήνες έχει μειωθεί σε λιγότερο από το μισό αυτή η διαδικασία. Ήταν σημαντικό λοιπόν, αυτά ήταν τα πιο επίμαχα σημεία προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα το ελεκτικό συνέδριο να δίδει τις εκθέσεις του ταχύτερα για να μπορούμε να αντιδράσουμε και εμείς ε, πιο γρήγορα. Βλέπω τον κύριο Γκάιερ. Θυμάμαι ότι αγωνιστήκαμε μέχρι την τελευταία στιγμή για τα θέματα αυτά. Γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Γκάιερ όλα τα επιχειρήματα που είχαν να κάνουν με τα θέματα της ε, απαλλαγής και πιστεύω ότι στην επόμενη μεταρρύθμιση ίσως θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά τα οποία δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν σε αυτόν, σε αυτόν τον τριγωνικό διάλογο αλλά έχουμε δώσει ένα αγώνα και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας ο οποίος στις πολύ δύσκολες αρχικές συνθήκες της ε, διαπραγμάτευσης έπαιξε ένα πάρα πολύ θετικό ε, ρόλο. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να είναι τόσο σε ένα πρόεδρο επιτροπής. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν γιατί μας βοήθησε σε την πολύ καλή ομαδική εργασία και ήταν πολύ καλό σημάδι ότι ήσασταν παρόν. Ε, ναι, ένα συνδευτικός ρόλος ουσιαστικά, διότι ήταν εξαιρετική η προεργασία που είχατε κάνει και σας αποτείω φορο τιμή, ε, κυρία Γκρέσλε. Ήταν μέγιστη η πρόκληση σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο και η έκβαση ε, φαινόταν δύσκολα προβλέψιμη στην αρχή. Με την αποφασιστικότητά σας όμως ε, ανταμυφθήκατε και σας συγχαίρω πραγματικά. χρησιμοποιήσαμε αυτό το παραθυράκι που υπάρχει για να τροποποιήσουμε το δημοσιονομικό μας κανονισμό. Σε μια πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έκριναν ότι ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής οι προτάσεις, όμως απεδείχθη ότι ήταν ιδιαίτερα πρόσφορες οι προτάσεις, οι οποίες καταλήξατε σε συνεργασία φυσικά με συναδέλφους. Σας συγχαίρω και πάλι θα χειροκροτήσουμε την εισηγητριά μας. Σχόλια. Ο κύριος Γκάια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση σε σχέση με την τροπολογία μου για τα πλεονάσματα του Αλικάντε, του Γραφείου Σημάτων στο Αλικάντε. Μπορεί να αγωνιστήκαμε ως το τέλος, αλλά ακόμα και αν δεν καταλήξαμε σε κάτι, είναι χρήσιμο να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει στη βάση ένα πρόβλημα. Πρόκειται για 500 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια και αυτό είναι κάτι το οποίο σωρεύεται σε σχέση με τον φορέα των σημάτων και με τη μείωση των ε, τελών για αυτών οι οποίοι διεκδικούν εμπορικά σήματα μπορεί να αυξηθεί το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να επιστραφεί στον προϋπολογισμό, δεν μπορεί να επιστραφεί στους πελάτες δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια λύση για το θέμα αυτό. Νομίζω στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δόθηκε, έγινε μια ψηφοφορία η οποία είναι πάρα πολύ τεχνικού χαρακτήρα και υπάρχει τώρα μετά από τον τρίλογο ένας διάβλος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα αυτά το πλεόνασμα της ε, υπηρεσίας ε, σημάτων ώστε οι εθνικές υπηρεσίες σημάτων οι οποίες ε, επομίζονται κόστος για να εφαρμόσουν ευρωπαϊκές αποφάσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα αυτά. Δεν είναι μονάχα λοιπόν μόνο μια επίθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά ουσιαστικά παίρνουν χρήματα οι εθνικέ υπηρεσίε για να εφαρμόσουν αποφάσει της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ε, ενέργεια την οποία δεν πρέπει να αποδεχτούμε. Ξαφνικά λένε οι εθνικές αρχές ότι εμείς για να εφαρμόσουμε τις ε, ευρωπαϊκές αποφάσεις χρειαζόμαστε κονδύλια. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το δεχτούμε γιατί θα χρησιμοποιηθεί αυτό το τέχνασμα και για άλλα θέματα. Υπήρξε λοιπόν αυτή η εξέλιξη στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εγώ τελείως τυχαία το έμαθα. Ήρθε ο σκιώδης εισηγητές μας από τους σοσιαλιστές σε μένα γιατί όλοι οι άλλοι θέλουν να το κλείσουν το θέμα αυτό χωρίς καθυστέρηση αλλά αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να επιληφθούμε και ενδεχομένω να έχουμε ένα ψήφισμα για να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή όλων στην Επιτροπή και ιδίως του Πρόεδρου μας. Ωραία τα περνάμε σήμερα το απόγευμα. Ε, αυτή η ιστορία ένα πράγμα μας δείχνει ότι είναι υπερβολική εκεί η κλίμακα που χρησιμοποιούμε ε, για τον υπολογισμό και πρέπει να μειωθεί. Οι εθνικές αρχές ανησυχούν δε διότι ε, θα είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια διατησία για αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, ε, άλλα σχόλια για αυτό το θέμα. Θα τα ξαναπούμε για τα σήματα. Και τώρα... Η έκθεση που όλοι περιμένανε, εκ των προτέρων, συγχαίρω το Χωζέ Μανουέλ. Ανέλπιστη νίκη, ένα δις. Αδύνατο, νόμιζαν όλοι. Εκείνος όμως καταφέρνει και τα αδύνατα. Ο κύριος Ντεπρέ φεύγει παρότι... Ε, κύριε Ντεπρέ, φεύγετε, αλλά αύριο θα μας πείτε για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, δεν έχετε κανένα επιπρόσθετο επιχείρημα. Ξέρω ότι σπαράζει η καρδιά σας, αλλά... Ε, κύριε Φερνάντες, μην νομίζετε ότι σας δίνουμε και λευκές επιταγές επειδή σας έχουμε τόσο τυφλά εμπιστοσύνη. Έτσι, προσοχή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εσάς, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, τους συντονιστές, που εξ αρχής με στήριξαν. Ευχαριστώ τους Σκιώδης, όλο το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, Κάνα μία δουλειά και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν αδύνατο. Όμως, να το τονίσουμε, δεν ασχοληθήκαμε μόνο με τη χρηματοδότηση. Και δεν το δημοσιοποιήσαμε, δεν κάναμε διαφήμιση, όμως αληθεύει καταφέραμε να έχουμε το ένα δις για να ε, μειώσουμε τις περικοπές αυτές που είχαν γίνει στον ορίζοντα 2020 και στο ΣΕΦ. Επίσης είχαμε πει ότι πρέπει στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και μέσα στον κανονισμό να συσταθεί το Ταμείο για τις Εγγύησεις Α, και να θυμίσω ότι τα 550 εκατομμύρια για το ΣΕΦ και τα 550 εκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 ε, καταφέραμε να έχουν μικρότερο αντίκτυπο. Δεν πειράξαμε τις γραμμές για τη θεμελιώδη έρευνα. Τα άρθρα 18 και 19 μεταφέρθηκαν ε, σε παράρτημα τα θέματα της διακυβέρνησης, αλλά το lifetime και ε, την αξιολόγηση την κάναμε εμείς. Εάν ε, είναι θετική αξιολόγηση θα συνεχιστεί η λειτουργία του Ταμείου. Εάν η ξεχωριστή, η ανεξάρτητη αξιολόγηση είναι μάλλον αρνητική, ε, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή νομοθετικού χαρακτήρα και το τρίτο σενάριο, αν είναι απολύτω αρνητική αξιολόγηση και δεν λειτουργεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να επιδιώξουμε την πάυση της λειτουργία του. Το πιο σημαντικό είναι η πλατφόρμα των συμβούλων για τις δημόσιες οντότητες είναι δωρεάν και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μόνο το 1 τρίτο. Αυτή η πλατφόρμα θα βοηθήσει και τις εθνικές πλατφόρμες ούτως ώστε να διασυνδεθούν και σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ε, οι επιτροπές τις καλύψαμε σχεδόν όλες. Ήτρε, τραν. Φτιάξαμε και τη δικτυακή πύλη για να προβάλλουμε τις επενδύσεις. Δώσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια στο Ταμείο αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πέραν αυτού, το Κοινοβούλιο θα παίρνει τις αρνητικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επενδύσεων με ρήτρα εμπιστευτικότητας, αλλά θα τις παίρνουμε τις αποφάσεις και για τις ε, θετικές αποφάσεις, αυτό που εγκρίνεται δηλαδή από το Συμβούλιο Επενδύσεων, αυτό που δεν απορρίπτεται, δημοσιοποιείται φυσικά. Έχει μια δημοκρατική νομιμοποίηση πλέον το Ταμείο. Μειώσαμε τον αντίκτυπο σε σημαντικά προγράμματα. Προσδώσαμε διαφάνεια, δημοκρατικό έλεγχο και όπως είπα, συμπεριλάβαμε τις προτάσεις των Επιτροπών, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που ήταν πολύ σημαντικές, τις προτάσεις ε, της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, επίσης στην πλατφόρμα μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο ε, Στατικών Επενδύσεων. έχουμε και ένα καινοτόμο μέσο που, συμπληρωματικό που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Φτιάξαμε το κείμενο διότι χρειάζεται ανάπτυξη η Ευρώπη και έχουμε ένα νέο εργαλείο για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι όλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την βοήθειά τους. Όλοι συνέβαλαν σε αυτό το θετικό ομολογουμένο αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάναμε και θα τη συνεχίσουμε σε όλες, ε, σε, όλα τα οικονομικά έτη. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ε, ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στον ορίζοντα 2020 ε, και στο ΣΕΦ επανέλαβα αυτή την πρόταση πολλές φορές και θα συνεχίσω να το κάνω. Α, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που καταφέραμε είναι ότι το Συμβουλίο ήθελε να δουλεύει επί τη βάση του προηγουμένου δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν ήθελε να μιλήσει για το μέσο ευελιξία, δεν ήθελε να μιλήσει για το άρθρο 14 και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, των συνολικών ε, περιθωρίων. Εμείς όμως θέλουμε να ε, εξακολουθήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για άλλα προγράμματα. Ήταν συλλογικό το έργο, ομαδική εργασία και σας ευχαριστώ όλους. Ε, εργάστηκαν εξαιρετικά όλοι. Και νομίζω μπορεί, να, μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπινους πόρους των πολιτικών μας ομάδων αλλά και της γραμματείας των Επιτροπών, κυρίως δε της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ όλους. Ça Αυτές είναι μεγάλες ε, ώρες. Είναι η τελική ευθεία. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Ποτέ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πνεύμα και το χιούμορ σου, Χωσέ Μανουέλ. Minimiser, minimiser l'impact <laughs> Αυτό που είπες, να ελαχιστοποιήσουμε, να να ελαχιστοποιήσουμε στο maximum τις επιπτώσεις. Ο, εντάξει, σοβαρά τώρα δεν ήταν τόσο εύκολο. Εγώ είμαι καινούριο στην Επιτροπή. Και όταν το Κοινοβούλιο δεν έχει αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ήμουν ποτέ υπουργό, αλλά ε, ως διπλωμάτης πάντοτε καμία εντολή. Και είναι κάτι σαν αυτιστικός ο διπλωμάτης. Δύσκολα τα πράγματα. Όμως χρειάζεται κανείς ταλέντο για να είναι εισηγητής. Για να προχωρεί η υπόθεση. Και να είναι όλοι καλυμμένοι για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η υπόθεση γιατί για να ελκύσουμε τους επενδυτέ χρειάζεται ένα γενικό πλαίσιο όσο γίνεται πιο αρμονικό, ήσυχο. Οπότε αν μπορέσουμε να βρούμε τώρα μια ισόρροπη απάντηση για την Ελλάδα αυτό θα είναι πολύ καλό γιατί πρόκειται για κάποια βεβαιότητα ε, που εδώ και εβδομάδες ε, επικρέμαται ε, για το πού θα καταλήξει το ελληνικό ζήτημα, αυτό δεν ήταν τόσο καλό για τις επενδύσεις. Είδατε, είδατε που ο κύριος Λετζέρη, εάν δεν μπορούν να ε, πληρώσουν οι Έλληνες τον σύνοριο φύλακα, αυτό είναι φοβερό πρόβλημα. Οπότε έτσι ανοίγει κερκόπορτα και η πύλη για την λάθρο μετανάστευση. Τέλο πάντων, επιτρέψτε μου αυτά τα σχόλια πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτη κυρία Γκάρδια Θάβαλ, ευχαριστώ Ευχαριστώ και εγώ θέλω να συγχαρώ τον, Χωσέ, τον Ζωζέ Μανουέλ και να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στον τριγωνικό διάλογο. Σαν εισηγητής μπόρεσε να διευθύνει θαυμάσια όλες τις διαπραγματεύσει και είχε φυσικά πλήρη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις θέσεις του. Ήταν δύσκολο το έργο του, ήδη και από το σχήμα του Τριλόγου, όπου ήταν 50 άτομα τα οποία διαπραγματευόντουσαν, παρά το γεγονός ότι υπήρχε χανεκπρόσωπη, υπήρχαν πολλές επιτροπές, πολλές πολιτικές ομάδες, ήταν σχεδόν σαν να είσαι στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όπως είπε ο πρώτος, κάποια στιγμή τελειώσαμε στις 8 το πρωί, πήγαμε να φάμε πρωινό και μετά πέσαμε να κοιμηθούμε. Και μόνο τότε μπόρεσαν να κλείσουν όλα αυτά. Είχαμε λοιπόν ένα τριγωνικό διάλογο, ο οποίος κράτησε 8-9 ώρες, γιατί τελικά ήταν όλες αυτές οι, οι δυσκολίες. Χρειαστήκαμε σχεδόν σαν 400 μήνυ συμφωνίες, την κάθε αιτιολογική σκέψη, την κάθε παράγραφο και αυτό κάναμε αυτό λοιπόν ήταν πολύ πιο πολύπλοκο από άλλους φυσιολογικούς τριλόγους. Είναι γενικά όμως αλήθεια ότι στους τριγωνικούς διαλόγους εμείς ως Κοινοβούλιο ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, δεν πρέπει να χάνουμε όμως ποτέ την ελπίδα και είναι και πολύ δύσκολη θέση της Προεδρίας γιατί κάθε φορά μετράνε αν θα μπορέσουν να έχουν πλειοψηφίες ή αν θα έχουν στο σβέρκο τους τις άλλες 27 χώρες οι οποίες θα τους πούν τι είναι αυτά που προτείνεται. Αυτό το σύστημα λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί με το χρόνο γιατί δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τρίλογο. Είδαμε ότι και με τη βοήθεια της Κομισιόν ακόμα που ήθελε να προχωρήσει το θέμα αυτό δεν έφτανε. Είχαμε το Συμβούλιο που ήταν απέναντί μας και αυτό έκανε πολύ δύσκολο το έργο του Κοινοβουλίου Νομίζω ότι αν ληφθούν όλα αυτά υπόψη, ήταν πολύ καλή η συμφωνία. Είχε πολλές προτάσεις στο Κοινοβούλιο. Είχαμε πολλούς τρόπους να βελτιώσουμε το κείμενο. Δεν ευδοκίμησαν όλες οι προτάσεις μας, αλλά νομίζω ότι το βελτιώσαμε αρκετά. Και αυτό φυσικά είναι το πρώτο τμήμα, τουλάχιστον από την πλευρά του, των προπολογισμών. Έχουμε πετύχει κάτι, έχουμε βελτιώσει την χρηματοδότηση. Αλλά αυτό είναι και τμήμα των διαπραγματεύσεων που θα πρέπει να κάνουμε για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου του 2017 και θα παίξει κάποιο ρόλο και στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι το πρόγευμα της ουσιαστικής τροποποίησης του δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να το σταθεροποιήσουμε αυτό και να διατηρήσουμε αυτό το επενδυτικό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και για το δικό σας ρόλο στις διαπραγματεύσεις, λέει ο πρόεδρος Σαρτουή, ιδίως εκείνο το βράδυ. Κύριε Μαραγάλ, και εσείς ήσασταν παρόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Πράγματι, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τόσο ενεργός όσο η κυρία Γουαρδέα Σαβάλ και ο κύριος Φερνάντες ίδιος, που προφανώς θέλω να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια μπορώ να εκφράσω κάποιες διαφοροποιημένες απόψεις με λιγότερο ενθουσιασμό από αυτά που είπαν οι εισηγητές και ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι βελτίωσε ουσιαστικά το αρχικό κείμενο της Κομισιόν και κατάφερε να ξεπεράσει την στάση εμπλοκής που το Συμβούλιο προέβαλε πάντα με πρόσχημα την ομοφωνία. Αλλά ας είμαστε σαφείς. Το κείμενο αυτό είναι σε κάποια απόσταση από αυτό που θέλαμε. Μπορεί ο καθένας να αποφασίσει πόσο μεγάλη είναι η απόσταση αυτή. Απέχει κάπως από το αρχικό κείμενο του Κοινοβουλίου. Και υπήρξαν κάποιες ε, <clears throat> ε αντιδράσεις από βουλευτές και από συγκεκριμένους βουλευτές που εκφράζανε κάποιες ε, αμφιβολίες, κάποιες ε, επιφυλάξεις για το τελικό αποτέλεσμα. Η πολιτική μας ομάδα θα συζητήσει αύριο το θέμα αυτό και υπάρχουν ε, προς όλες τις κατευθύνσεις επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε από τις τρεις επιλογές και φυσικά μεταξύ αυτών είναι και η θετική ψήφος. Θα ακούσουμε όμως όλες τις απόψεις οι οποίες ε, πρέπει να τύχουν σεβασμού σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων της Ευρώπης 2022 και του Connecting Europe Facility. Βλέπουμε ότι μειώνονται πάρα πολλοί προγράμματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με την έρευνα κτλ. Ενώ διατηρούνται όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με συμφωνίες με μεγάλους, μεγάλες διεθνείς εταιρείες, ξέρουμε ότι αυτό είναι μια παράδοση. Δεν Και αναγκαστήκαμε επίση να δεχτούμε και είναι επιτυχία ότι διατηρήθηκε αυτό το δισεκατομμύριο στον προϋπολογισμό, αλλά χρειάστηκε να απαρτηθούμε τη χρήση των περιθωρίων και την ε, έννοια της μεταρρύθμισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και για τα θέματα της ευκυβερνησίας, της διακυβέρνησης, πρέπει να κρίνουμε θετικά ορισμένα πράγματα. Στο τομέα της αιρεσιμότητας, υπήρξε κάτι θετικό σε σχέση με την έννοια του βαθμολογίου. Αυτό ήταν θετικό που έγινε δεκτό, παρά το γεγονός ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα οποία προβλέπονται από την Κομισιόν και πρέπει να εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε πως, πολλές, πως προς πολλές κατευθύνσεις το αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν πραγματικά συναρπαστική η διαπραγμάτευση. Δεν μπόρεσα να ήμουν στο τέλος αυτής της διαδικασίας όπως είπε η κυρία Γουάρδα Σαμπάλ εγώ είχα φύγει από την Ευρώπη τότε ήμουν στην Παλαιστίνη Εν πάση περιπτώσει αύριο θα έχουμε τον τελικό λόγο για το θέμα αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απαραίτητες αποχρώσεις και τα σχόλιά μας για το θέμα αυτό ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω κύριε Πρόεδρε. Αυτό ξεκίνησε ως ένα σχέδιο, ένα συγκεκριμένο σχέδιο με στόχους ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας την κρίση στην οικονομία μας και την κοινωνική ε, δυσχέρεια στην Ευρώπη, αλλά γίνεται πια ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και όχι ένα σχέδιο που υπάρχει θέληση από πολλούς να πάρει μόνιμο χαρακτήρα, είναι μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης, έναντι του αρχικού σχεδίου που είχαμε στα χέρια μας. Και στην περίπτωση αυτή, όπως έλεγε η κυρία Γουέρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό και σε οποιαδήποτε διαδικασία ε, ελέγχου και αναθεώρησης του Ταμείου θα πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι για να ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να δεχτούμε ή όχι αυτά που προτείνονται και κατά πόσο συνάδουν με τους αρχικούς στόχους αυτού του σχεδίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ε, επιδοκιμασία μου για το τελικό αποτέλεσμα που είναι πολύ καλύτερο από το αρχικό κείμενο Ακόμα και τα σημεία που δεν πέρασαν δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι επισκιάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Στην κοινή συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ ε, είπαν ορισμένοι ότι το αποτέλεσμα μπορεί να ε, δικαιολογήσει και την όλη διαδικασία. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, πάντως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην επαναληφθώ αυτά που έχουν γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Είχαμε μια κοινή επιτροπή, λέει ο πρόεδρος. Ε, είναι μια, ένα κοινό, μια κοινή στιγμή ευτυχία, α το πω έτσι. Έτσι προετοιμάζουμε την, ε, το δυνατόν μέγιστη συσπήρωση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, καλά δεν τα λέω. Έχουμε και κάτι λεπτομέρειες, ε, π.χ τη σύμβαση ε, ανάμεσα στην Επιτροπή και την ΕΤΕ θα γίνουν ακόμη ε, πολλές συσκέψεις. Ήταν τόσο μεγάλη η ευτυχία και ο ενθουσιασμός στις κοινέ συνεδριάσεις που θα το παρατείνουμε. Ε, και εσύ Γιατί έχουμε το σχέδιο σύμβασης και εμείς θα γνωμοδοτήσουμε γι' αυτό. Ε, και πρέπει να ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και πλειοψηφία για να υπερψηφιστεί το κείμενο. Εάν ε, παραμένουν ε, σκεπτικοί και έχουν ενδιασμού οι συνάδελφοι, τώρα είναι η σωστή στιγμή να προσπαθήσετε με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή σας να τους μεταπίσετε. Όμως επειδή πρέπει να πρεσβεύει η εμπιστοσύνη, μην ξεχνάμε ότι δεν χρησιμεύει τίποτα απολύτως αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Για να καταδείξουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη μας. Έχουμε ήδη εμείς υποθέσει ότι θα υπερψηφιστεί αύριο το κείμενο και έχουμε ήδη οργανώσει το κοκτέιλ μετά την επιτυχία έκβαση της ψηφοφορίας. Αχα, τι νομίζατε. Και σας προσκαλώ. Όπως και να, το ε, να ψηφίσετε αύριο, σας προσκαλώ. Είναι για να δείξουμε την ε, ευχαριστησή μας ε, και να συγχαρούμε όλους όσους κατήσαν δυνατή αυτή τη τόσο θετική έκβαση του τριλόγου. Ε, Μανουέλ σήμερα το πρωί μας έλεγες πώς μπορεί κάποιος να βρει προστιθέμενη αξία στα ευρωπαϊκά κονδύλια, γενικότερες κρατικές δαπάνες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αποδεδειγμένα προστιθέμενη αξία. Και ξαναλέω, από τι οφόρο τιμή στον εισηγητή, στους κοιόδης, σε όλους όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή των εργασιών. Εγώ είμαι σχετικά καινούριο και πραγματικά βλέπω πόσο μεγάλη είναι η πραγματογνωμοσύνη αλλά και η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων ε, είναι εξαιρετικά ποιοτική συνεργασία και ξαναλέω ότι ε, είναι ε, αξιοθαύμαστη η πραγματογνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω διότι ειδικά κατά τις 7 το πρωί εκεί στον τελευταίο τρίλογο που έγινε Αναρωτιόμασταν όλοι οδηγεί κάπου αυτό, διότι ακόμη και σε επίπεδο ανθρωπίνων επαφών, ε, ψυχολογικών αντιδράσεων, ε, νεύρων, νευρικής φόρτισης, ε, ήταν αρκετά βάρια η διαδικασία και τελικά το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί και ήταν τελικά θετικό το αποτέλεσμα, θα ήταν και κρίμα να, θυσιαστούν, ε, θυσιαστεί τόσο ιδρώντας και τόσες ώρες, τόση ενέργεια χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ελπίζουμε τα καλύτερα για αύριο και τι ώρα είναι, 7-8, τι ώρα είναι το κοκτέιλ. Στις 8. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική αυτή η περιπέτεια και σας ευχαριστώ. Για να δούμε αν θα λειτουργήσει. Πρέπει δηλαδή αυτός ο μηχανισμός που φτιάξαμε να είναι αποτελεσματικός και για να αποφασίσουν οι ιδιώτες επενδυτές να διατρέξουν τον κίνδυνο με αυτήν την υπέροχη εγγύηση που τους δίνουμε. Μόχλευση 15 δεν είναι αμεληταίο. Χρειάζεται όμως και ε, κατάλληλα προσαρμοσμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη ολοκλήρωση ενίας αγοράς, ο κατακαιρματισμός παραμένει μεγάλος και σίγουρα αυτό είναι δυσίωνο για τις ιδιωτικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι θα δείξουμε όλη την ίδια ενέργεια για να προωθήσουμε με τη σειρά, την, ε, με τη σειρά της, συγγνώμη, την ενιαία αγορά για να ε, άρουμε όλους αυτούς τους φραγμούς και προσκόμματα προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης θα είναι μεγάλη προσταμένη έξια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τουλάχιστον το 20% αυτού του κονδυλίου θα διοχετευτεί άμεσα. Ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι οποίες παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας. Είδου, πλησιάζουν και οι διακοπές και μην ξεχνάμε ότι είχαν επιτυχή έκβαση τρεις τριλογοί για τις πληρωμές. Ε, υπάρχουν κάποιοι που έχουν ακόμη τις αμφιβολίες τους, αλλά το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε ήδη σήμερα το πρωί ότι είχαμε επιτυχία. Το, ο τρίλογος ε, για τις ε, ε, ε, πληρωμές, ε, χάρη κυρίως στην αποφασιστικότητα της κυρίας Γκρέσλεμ και για το ΕΦΣΙ, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, πολύ καλό το αποτέλεσμα γιατί υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ε, τσαμπουκαλευόμενοι, θα το έλεγα έτσι, ε, δεν πρέπει να κουμπίσετε, τολμήσετε να κουμπίσετε το ΣΕΦ και τον ορίζοντα 2020 και ο Χωζέ Μανουέλα έψαχνε κακομύρης να δει πώς μπορεί να βρει λογικά επιχειρήματα και μπόρεσε τελικά ούτε που ξέρω πώς να ε, ξεκλέψει ένα δις ολόκληρο. Πραγματικά καταπληκτικές οι επιδόσεις σου και η αποφασιστικότητα που έδειξες και ήσουν και αποτελεσματικός και κόμψος ε, στα διαβήματά σου. Λοιπόν, νομίζω αρκετά. Ήταν ιδιαίτερα φορτωμένη η μερίσια διάταξη. Η μέρα ήταν πολύ φορτωμένη. Από τις 9 είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Για τη συνεδρία της Επιτροπής και το βράδυ στο κοκτέιλ.